Αγαπητοί μου συνάδελφοι, άρχεται η ακρόαση με τριπλή προεδρία, διότι εκτός από την Επιτροπή Προπολογισμών συμμετέχουν και η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, καθώς επίσης και η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, αντιπρόεδρο προτινόμενη. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι το παράρτημα 16 του κανονισμού μας, το Κοινοβούλιο αξιολογεί τους προτινόμενους επιτρόπους επί τη βάση της επάρκειάς τους, της γενικότερης δηλαδή, της ευρωπαϊκής τους προσήλωσης και της προσωπικής τους ανεξαρτησίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης αξιολογεί τη γνώση του ενδεχομένου χαρτοφυλακίου, καθώς επίσης και τις επικοινωνιακές του ικανότητες. Θα ήθελα να θυμίσω ότι πριν από την ακρόαση η αντιπρόεδρος ε, που προτείνεται έχει ε, απαντήσει γραπτό σε ένα προπαρασκευαστικό ερωτηματολόγιο. Οι βουλευτές έχουν λάβει τις γραπτές απαντήσεις σε όλες τις γλώσσες. Η συζήτησή μας θα διαρθρωθεί ως εξής η προτινόμενη αντιπρόεδρος θα κάνει μια πρώτη προφορική εισαγωγή που δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει τα 15 λεπτά και στη συνέχεια στο τέλος της ακρόασης θα έχει και 5 λεπτά στη διάθεσή της για να δευτερολογήσει και να κλείσει. Μετά τα εισαγωγικά σχόλια θα γίνει η ακρόαση με 45 ερωτήσεις των βουλευτών, στις οποίες θα απαντά άμεσα η προτινόμενη αντιπρόεδρος. Τρία λεπτά είναι το σύνολο, ένα λεπτό για την ερώτηση και δύο λεπτά για την απάντηση. Ο πρώτος γύρος ερωτήσεων αφορά ένα πρόσωπο από κάθε πολιτική ομάδα. Ο δεύτερος γύρος θα είναι σε τρεις ενότητες, ανάλογα με τις τρεις επιτροπές που συμμετέχουν με την εξή σειρά. Πρώτα, θα ρωτήσουν οι συνάδελφοι της Επιτροπής Προϋπολογισμού, στη συνέχεια ε, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τέλος των νομικών θεμάτων. Θα ήθελα επίσης να σας επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι έχουμε δύο ερμηνεία σε 22 γλώσσες. Όλοι οι βουλευτές λοιπόν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη μητρική τους γλώσσα. Παρακαλούνται όμως οι ομιλητές να λαμβάνουν υπόψη ότι θα μεταφράζονται αναγκαστικά τα όσα λέγουν, οπότε δεν θα πρέπει να μιλούν πολύ γρήγορα για να μπορούν να μεταφράζονται. Επίσης, η συνεδρίαση μεταδίδεται απευθείας ε, στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Επίσης, μαγνητοσκοπείται και θα είναι στη διάθεσή σας πάντα στην ίδια ιστοσελίδα. Πριν δώσω το λόγο στους δύο συναδέλφους, πρώτα στη συνάδελφο της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού και στη συνέχεια στον κύριο Σφόποντα. Κυρία προτινόμενη Αντιπρόεδρε, με προσοχή παρακολουθούμε την κατάρτιση του προπολογισμού για το 2015. Υπάρχουν πάρα πολλές ε, εκκρεμότητες για πληρωμές, outstanding payments και περιμένουμε μια διορθωτική απάντηση για να λυθεί αυτό το θέμα και να εξασφαλίσουμε ε, αυτό το θέμα και να μην υπάρχει ένα έτσι, ύπουλο υποχθώνιο χρέος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 2016 ε, έχουμε και το πολιετές πλαίσιο, θα ασχοληθούμε το 2015 όμως με αυτό επίσης και προσέχουμε πάρα πολύ και παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς ε, το μέλλον των 300 δισεκατομμυρίων που εξήγηλε ο κύριος Γιόγκερ για το 2015 και επέκεινα. Επίσης παρακολουθούμε και μας ενδιαφέρει να δούμε πώς θα διαμορφώσετε και τι θα προτείνετε για τους ιδίους πόρους για να μπορεί το Κοινοβούλιο να ψηφίζει κάποια στιγμή τη φορολογία και να μας δώσετε και ένα όραμα, μια θεώρηση για το πώς αντιλαμβάνεστε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της Ευρωζώνης και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Θα δώσω τώρα μέσω στο λόγο στην κυρία Ίγκεμπορ Γκρέσλε, πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του Προβολογισμού. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ συνάδελφε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω θερμότατα την Επίτροπο κυρία Γεωργιέβα, εξ ονόματος και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Έχουμε νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή με νέα χαρτοφυλάκια. Ε, πριν το 2004 είχαμε αντίστοιχη κατανομή με τη σημερινή. Βλέπουμε ευκαιρία σε αυτή τη νέα κατανομή για τον προϋπολογισμό, τον έλεγχο του προϋπολογισμού και την καταπολέμηση της απάτης στα ίδια χέρια. Πάνω από 5.000 ε, υπαλλήλους έχετε, ένα έβδομο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό την άμεση δικαιοδοσία σας, οπότε είστε ε, και η μόνη αντιπρόεδρος που έχετε ε, άμεση σχέση με τη γραφειοκρατική, τη διοικητική μηχανή. Γενικά βλέπουμε ως ευκαιρία ε, τη νέα κατανομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα χαρτοφυλάκια. Χαιρόμαστε για την ανταλλαγή απόψε. 14 από τις 45 ερωτήσεις αφορούν ε, ζητήματα της δικής μας αρμοδιότητας Επιτροπής Ελέγχου και εκεί θα έχουμε τη διαδικασία αυτή του ping pong, τρία λεπτά, στην αρχή εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων και μετά ε, μεμονωμένοι βουλευτές. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας προς όφελος και συμφέρον των φορολογουμένων ανδρών και γυναικών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. La parole à Pavel Svoboda, président πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα κυρία Γεωργιέβα. Καλώς ήρθατε σε αυτή την ε, ακρόαση. Ε, σας ευχόμαστε από πλευρά τη Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, τη Επιτροπής της οποίας ε, προεδρεύω. Εμείς σας έχουμε απευθύνει ένα συγκεκριμένο περιορισμένο αριθμό ερωτήσεων για σήμερα. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, γιατί σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι σημαντικός ο προηγουμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ορθή του εκτέλεση είναι μια μέρημνά μας, είναι κάτι που μας καίει και να δούμε τον προπολογισμό το Κοινοβούλιο είναι πεπισμένο σημαίνει ότι είναι κορυφαία σημασία, ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε επιτυχή εκτέλεση, να έχουμε εποπτεία των προγραμμάτων των πολιτικών και να γίνονται όλα αυτά για το συμφέρον, για το καλό των πολιτών, των Ευρωπαίων, των επιχειρήσεων και έτσι οι περιφερειακές υπηρεσίες, οι οργανισμοί, τα θεσμικά όργανα, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να ε, υπολογίζει σε κάποιους άνδρες αλλά και γυναίκες οι οποίοι να έχουν τις, ε, ε, τα κίνητρα, να έχουν τη θέληση, να έχουν τις δεξιότητες και τα προσόντα. Εσείς θα έχετε όπως έγινε ο κύριος Γιούνκερ τις ανθρώπινους πόρους, επομένως θα ασχοληθεί με την κινητικότητα, ε, με το προσωπικό άμεσα αλλά και έμεσα και για κάποια άλλα πάρα πολύ σημαντικά θέματα για το προσωπικό σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, υπηρεσίες και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είσαστε η αρμοδία για την εύρυθμη λειτουργία των ανθρώπων παράγοντας στην Ένωση. Εμείς έχουμε υπόψη του πόσο σημαντικό είναι το καθήκον σας και πόσο θα πρέπει το προσωπικό ε, να συμμετάσχει και θα πρέπει και εμείς να συμμετάσχουμε σε αυτή τη διαδικασία εξίσου με τις άλλες δύο συνομόδιες επιτροπές και περιμένουμε να ακούσουμε την ενακτήρια εισήγησή σας. Ο Πρόεδρος, Αρτή. Κύριε Υποψηφία, Αντιπρόεδρε, έχετε το λόγο.